Πάρα πολύ μεγάλη. Pardon, madame, pardon, madame, oui, puis après, monsieur le rapporteur concurrent. Ähm, Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte jetzt nur noch mal, weil ich das so ungeheuer spannend finde, dass auf... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ σαφή ερώτηση του συναδέλφου Γκρέσλε. Ça marche German is an unknown uh, language. Ακούνε καλά τα ελληνικά παρακαλώ. Ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ. Ich wollte nur auf die... Θα ήθελα, λέω, να απαντήσω στην πολύ ακριβή ερώτηση που υπέβαλε η συνάδελφος Γκρέσλε ε, και να υποβάλω μια συμπληρωματική ερώτηση. Ερωτήθη Ποιε είναι οι πληρωμές που κατευρύθησαν 21 31η 8 2009 στο Κοσοντόι. Ακούσαμε έτσι πολύ ε, εφραδείς απαντήσεις, αλλά δεν ακούσαμε το ποσό ακριβώς. Αυτό θα ήθελα και εγώ να το ακούσω. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Διευθυντά, μπορείτε να δώσετε το στοιχείο αυτό γραπτά. Γραπτά, ωραία. Θα σας ε, μεταβιβαστούν πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Ωραία. Θαυμάσια. Αλλιώς θα βασανιστεί ο κύριος Γενικός Διευθυντής. Ο κύριος Γενικός Εισηγητής τώρα παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε. <clears throat> Mr. Chairman, I have to recognize that we are... Πρόεδρε, αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε πια στη συνέδρια κλεισμένων των θυρών και γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με υποστήριξαν κατά διάρκεια της συζήτησης. Και τώρα έχουμε ένα μήνυμα προς όλους, ιδίως στο Συμβούλιο, ότι η Επιτροπή μας εδώ υποστηρίζει τα αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης. και ε, από την άλλη μεριά έχουμε τη δύσκολη κατάσταση για τον πρόεδρο του Συμβουλίου και θα πρέπει να δούμε πού θα γίνουν οι θυσίες κατά τη διάρκεια της Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, ότι η συζήτηση για το Κοσλοτούι δεν είναι συζήτηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλγαρίας και ούτε λέγεται ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα που χρειάζονται. Υποστηρίζουμε την ιδέα, υποστηρίζουμε το πλήσιμο. η συζήτηση γίνεται μόνο για τα μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι ο τίτλος που προτείνει η Κομισιόν είναι ο ιδανικότερος. Δεν θα μας οδηγήσει την καλύτερη δυνατή λύση. Και πιστεύω ότι η πρόταση που έχουμε τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η χρηματοδότηση να αποστείλουμε δηλαδή ένα κοινό μήνυμα από το Κοινοβούλιο, να αρχίσουμε τη χρηματοδότηση αυτή ευέλικτα. Δεν είναι υπόσχεση ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες ευελιξίας επί τέσσερα χρόνια. Ήταν κάτι τέτοιο. Εγώ υποστηρίζω τις επικρίσεις για την λογική αυτή. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι είναι δυνατόν να επιληθεί. Άκουσα πάρα πολλά ενδιαφέροντα από την Κομισιόν και χρειάζομαι ε, κάποιες προσωπικές συζητήσεις ίσως ε, για κάποια από αυτά τα σημεία. ή σήμερα ή μετά ή αύριο για να είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα σωστά γιατί ορισμένα που άκουσα με εξέπληξαν. Από την άλλη μεριά θα προσπαθήσω να καταλάβω αυτά που άκουσα. Αυτά σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά, ευχαριστώ όλους τους συνάδελφους και τον ε, Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής. Νομίζω ότι μπορέσαμε κατά τη διάρκεια των ε, δύο αυτών ωρών να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων που θα είναι πολύ χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην μεθαυρινή συνδιαλλαγή. Μια παρατήρηση μόνο, μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το Κοσλοντούι. Προσωπικά το μάθημα, το δίδαγμα που αποκαμίζω από αυτό το πρόβλημα και από αυτή την εμπειρία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις νομικές βάσεις, ώστε να μην επιβάλλουμε στους εαυτούς μας άχρηστες περιορισμούς από τη στιγμή που θέλουμε να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει και να ενεργήσει γρήγορα. Ο στόχος του σχεδίου ανάκαμψης ιστορικά Plan ήταν να μπορούμε να ενεργήσουμε γρήγορα, να περάσουμε ε, συμβάσεις ε, γρήγορα για να μπορέσουμε να, ξεκι... να, να προωθήσουμε την οικονομία και γρήγορα ναι, ε, ενέργειες νέου είδους και καθαρή ενέργεια. Αν το είχαμε φτιάξει λιγότερο συγκεκριμένα και με ευρύτερη φάση, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι το να κλείσουμε το Κοσλοντούι και την παλιά, τον παλιό σταθμό του Κοσλοντούι να μην μπορεί πλέον να βλάψει ώστε να στραφεί η παραγωγή ηλεκτρισμού στη Βουλγαρία προς την νέα ασφαλή ενέργεια να είναι όλα αυτά μέσα στο πνεύμα του σχεδίου ανάκαμψη. Όμω η νομική βάση δεν συντάχθηκε με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό και χρειάζεται να κάνουμε αυτέ τι δημοσιονομικέ ακροβασίε. Προτίζω τώρα να περάσουμε στον χρόνο εργασία και αφού έχουμε το... η τιμή να έχουμε μαζί μα τον Αλέχο Βιτάλ Κουάντρα, τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνο για την ε, πολιτική την κτηριακή αλλά και για τον προπολογισμό. Ζήτω συγγνώμη καταρχήν για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση και δύσκολη συζήτηση και να μην τον καθυστερήσουμε περισσότερο. Να περάσουμε άμεσα λοιπόν στο σημείο 9 τη ημερησίας διατάξεω, δηλαδή το σχέδιο τα σχέδια μεταφορών ε, για τα άλλα τμήματα. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Λεβαντόφσικη και να ξεκινήσουμε από το σε 17 που αφορά το Κοινοβούλιο και επί το οποίο ο κύριος Λεβαντόφσκι και ο κύριος Μπουκρός θα λάβουν το λόγο. Thank you. Uh, before, before... Σας ευχαριστώ. Πριν να μπούμε στα βαρέα βάρη που είναι το 17, να κάνω μια παρατήρηση για το 21 που αποσύρθηκε και που ήταν τμήμα της αντιπαράθεσής μας στην τελευταία συνεδρίαση ε, όπου πρόκειται για τη διοργάνωση συνεδριάσεων ανωνύμων πολιτικών ομάδων χωρίς χρήματα. Φαίνεται πως επιπλέον αυτές οι συνεδριάσεις έχουν ακυρωθεί, άρα μπορούμε να ακυρώσουμε και αυτό το αντιφατικό, την αντιφατική μεταφορά, την 21. Δεν χρειάζονται κονδύλια γιατί η ομάδα εγκατέλειψε τις επιπλέον ε, συνεδριάσεις. Έχουμε λοιπόν το σε 17 τώρα. Όσον αφορά την πολιτική στρατηγική, είναι ξεκάθαρη και ο κύριος Κάτρας μπορεί να την επιβεβαιώσει. Έχουμε το πράσινο φως από το Προεδρείο για την αγορά επιπλέον χώρου για το Κοινοβούλιο. Έχουμε και το πράσινο φως όσον αφορά την χρηματοπιστωτική προσφορά. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα μίσθωσης με, με προτίμηση για αγορά. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2011. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην καθαρά δημοσιονομική πτυχή ε, όταν λέμε καθαρά δημοσιονομική πτυχή ε, σημαίνει πως ε, στόχος είναι εμείς πολιτική έχουμε να αγοράζουμε και όχι να νοικιάζουμε για να μπορούμε να περιορίζουμε το δημοσιονομικό βάρος στο μέλλον αλλά υπάρχουν και οι άλλες πτυχές της απόφασης και νομίζω πως και οι παρατηρήσεις του κυρίου Μπούκρου θα πρέπει να είναι σχετικές με το θέμα. Θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο πλαίσιο της γενικής κτηριακής στρατηγικής μας και όχι στρατηγική αναπερίπτωση. Ε, και γι' αυτό Νομίζω πως θα πρέπει να συζητήσουν, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την αγορά του κτηρίου ΤΡΕΦ 1. Θέλετε να μιλήσετε τώρα κύριε Βιταλκού ή μετά τον κύριο Μπουτουκρός. Νομίζω πως ίσως είναι καλύτερο να ακούσουμε τον βουλευτή της Επιτροπής Προπολογισμού. Ο κύριος Μπουκρός λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον σπουδαίο μου φίλο Γιάννους Λεβαντόφσκι πως ε, φυσικά τα δημοσιονομικά θέματα είναι αλληλένδετα με τα μη δημοσιονομικά. Ωστόσο, τμήμα της σύστασής μου επίσης αναφέρεται στην, ε, στα, στα οικονομικά, όχι μόνο στο κτίριο. Όπως έχω στείλει και λέω μάλλον και στην επιστολή που έχω στείλει σε κάθε ε, βουλευτή της Επιτροπής, μετά από εκτεταμένες έρευνε. Ε, μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή Προπολογισμού μπορεί να λάβει θετική απόφαση επί της αρχής. Πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει ή όχι την δημοσιονομική μεταφορά σε αυτό θα επανέλθω όταν θα μιλήσουμε για τα χρηματοδότηση, για τα οικονομικά. Αλλά υπάρχουν κάποια εκρεμή ζητήματα. Να αναφέρω τα εξή τρία που θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω και που μπορεί να ρυθμιστούν καλή την πίστη πολύ σύντομα. Και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτή τη συναλλαγή. Βεβαίω η απόφαση επί της αρχής μπορεί να βασιστεί σε δύο σημαντικούς τομείς. Ένας είναι και δεν θέλω να μακρηγορήσω από αυτού. Όλοι γνωρίζουμε γιατί χρειάζεται περισσότερο χώρος. Το άλλο είναι η εξαιρετικά ευνοϊκή τοποθεσία του κτηρίου, δηλαδή ακριβώς δίπλα στη, σε αυτές εδώ τις εγκαταστάσεις, σε αυτές, αυτά εδώ τα κτίρια. Ένα σημαντικό στοιχείο, παρακαλώ να με προσέξετε αυτό που θα σας πω, είναι ότι πρόκειται για το μισό ενός μεγάλου κτηρίου και το άλλο ήμιση επίσης θα βγει προσπόληση πολύ σύντομα. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί Μπορεί να μπορούμε να αγοράσουμε και τα δύο κομμάτια του ιδιοκτηρίου σε πολύ καλή τιμή και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να περιμένουμε για λίγο. Γιατί όπως σας είπα μπορεί να βγει προσπόληση και το άλλο κομμάτι. Ίσως θα ήταν λοιπόν πιο καλή η τιμή αν αγοράζαμε και τα δύο. So, ε, ε, very important. Ε, last time when... Κάτι ακόμα που ήταν σημαντικό την περασμένη φορά που το συζητήσαμε μίλησα για το θέμα του αμίαντου που είναι ιδιαίτερα προσφυλές στους πράσινους αλλά και προσφυλές σε όλους μας. Τώρα μετά από πιέσεις επιπιέσεων προς την διοίκηση τελικά την Παρασκευή το απόγευμα, που δεν είναι και πολύ καλή στιγμή, λάβαμε ένα έγγραφο στα φλαμαδικά 17 σελίδων το οποίο διαβάσαμε, διαβάσαμε όσο και αν σας κάνει εντύπωση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ανακαλύψαμε ότι το κτίριο περιέχει αμύαντο. Επιτέλους το αναγνώρισαν αυτοί που έκαναν την προηγούμενο έλεγχο, αν και είναι αρκετά περίπλοκο. Λέει ότι οι σωλήνες ε, και τα διάφορα στοιχεία είναι τμήματα από τα οποία μπορεί να αφαιρεθεί ο αμύαντος, αλλά από ό,τι φαίνεται αμύαντος υπάρχει και στη δομή του κτηρίου, πράγμα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα προβληματάκι εδώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν και τα πιστοποιητικά λένε ότι η συγκέντρωση ινών αμοιάντου στον αέρα είναι κάτω από το επίπεδο χιλίων ανακυβικό μέτρο που είναι το πρότυπο για τα θέματα υγείας, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο ίδιο έγγραφο πως ετησίως θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Ω προς αυτό πιστεύω πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιορίσει το πρόβλημα. Οποτεδήποτε δηλαδή το επίπεδο αμοιάντου ξεπερνά αυτό το κατόφλι, που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως ε, όριο για την ανθρώπινη υγεία, θα πρέπει να επιβάλλεται μία εκαθάριση καθώς ε, και θα υπάρχει περισσότερο κόστος γιατί θα πρέπει να μετακινηθούν αυτοί που θα εργάζονται εκεί. Αυτά. Ε, λοιπόν, για τον αμύαντο και πραγματικά την επόμενη φορά φροντίστε να μας στείλετε τα έγγραφα σε άλλες εξωτικές γλώσσες. για να μπορέσουν να μετακινηθούν εκεί οι βουλευτές μαζί με το προσωπικό τους θα πρέπει να γίνουν περισσότερα έργα. Αν όμως μετακινηθεί τμήμα της διοίκησης εκεί δεν χρειάζεται κανένα έργο να γίνει γιατί το ίδιο το κτίριο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο. Και επίσης υπάρχουν οικονομικές συνέπειες, συντηρήση και γενικό κόστος λειτουργίας. Τέλος, να έρθω στο θέμα της χρηματοδότησης, που είναι επίσης σημαντικό για μένα. Διότι δεν συμφωνώ απαραίτητο, αλλά κατανοώ την παρατήρηση που έγινε και ότι τώρα είναι πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν έχω καταλάβει καλά, να αγοράζει και να μην νοικιάζει τα κτίρια του. Εντάξει, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό, να το αμφισβητήσω, αλλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη πρώτον ότι η βελγική κυβέρνηση μαχαιροστά χρωστά 7 εκατομμύρια λόγω της 70 ε, εκατομμύρια, 70 όχι 7, 70 εκατομμύρια λόγω της ανακατασκευής ολόκληρης της πλατείας Λουξεμβούργου. Δεν το έχω δει ποτέ γραπτός, αλλά κάπου υπάρχει. Όταν δηλαδή θα πρέπει να δούμε ξανά ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δούμε το ισοζύγιο και όχι τον ετήσιο προπολογισμό. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα απαιτήσουμε από τη βελγική κυβέρνηση. Τώρα, Αν το κάνουμε αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε leasing και, και με επιλογή αγοράς, δεν χρειάζεται να γίνει τόσο περίπλοκη υπόθεση, θα μπορούμε να τα αγοράσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση και γι' αυτό και θεωρώ πως είναι σημαντικό η Επιτροπή μας τουλάχιστον να το γνωρίζει. Εν γέννη, θα έλεγα ότι είμαι υπέρ Euh, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Ευχαριστούμε για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε από τότε που ξεκίνησε αυτό το θέμα. Τώρα πριν ο κύριος Αντιπρόεδρος λάβει τον ε, λόγο, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και στην περασμένη συνεδρία τη Επιτροπή είχα ζητήσει το λόγο για το θέμα αυτό. Και θα το ξανακάνω. προτιμά να αγοράσει από το να νοικιάσει το κοινοβούλιο. Αυτή η γραμμή είναι λογική, εφόσον οι τιμές ανεβαίνουν στην αγορά των ακινήτων. Όταν είναι στις σημεία όμως υπέφτουν οι τιμές, δεν είναι πολύ λογική αυτή η στρατηγική. Και αν δεν έχουμε καλύτερα επιχειρήματα για την αγορά από το «το κάναμε πάντα έτσι», δεν θα προστατευτούμε από κακή ποιε επενδύσει. Στην άλλη γωνία από το Τρέβενα υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο γραφείων με μια μεγάλη ταμπέλα ότι νοικιάζονται πάρα πολλά γραφεία συγκεκριμένου και πάρκινγκ. Όταν λέμε ότι έχουμε 125 περισσότερες ε, ε, θέσεις απασχόλησης μετά από κάθε διεύρυνση, θα μπορούμε νομίζω με την προβλεπόμενη διεύρυνση που θα έχουμε 250 ε, υπαλλήλους περισσότερους, να βρούμε κάποια δυνατότητα που να μπορούν πραγματικά να αντέξουν έστω να περνάνε την άλλη μεριά της ε, Ρουμπελιά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ καλή επιλογή το να αγοράσουμε. Δεύτερον, αμύαντος. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά παίρνουν την υγεία των εργαζομένων οι συνδικαλικές εκπροσωπήσει του σώματο. Αλλά από την προσβέρνη μου εργασία ξέρω ότι το αμύαντος αποτελεί μία ε, απειλή της υγείας των εργαζομένων. Γιατί οι ίνες αμοιάντου ξέρουμε ότι οδηγούν στην δημιουργία καρκίνου του πνεύμονα. Εάν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στο κτίριο Τρεβένα, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου αυτοί που θα εργαστούν σε αυτό το κτίριο να μην απειληθούν α, όσον αφορά την υγεία τους. Αν δεν μπορεί να υπάρχει οριστική λύση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και μη νομίζω, γιατί θα πρέπει τότε να κάνουμε μια ανακαίνιση για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή της υγείας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λοιπόν στην αγορά, στην τιμή της αγοράς. Εγώ δεν θα ψηφίσω αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να συζητήσω και στα μέλη της ομάδας μου να απασχόλω τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιπρόεδρος. Έχει το λόγο. Uh, thank you, thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής των Προπολογισμών για την τόσο αξιολογική γνώμη τους για το θέμα μας. Όπως γνωρίζετε, πιέζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πιέζει για περισσότερο χώρο για πολλούς λόγους. Με δεδομένη συνήθεια της Λισαβόνας είμαστε αναγκασμένοι να αυξήσουμε το προσωπικό. αλλά και ελαφρώς τον αριθμό των βουλευτών. Πρώτη τι αυτή, η δεύτερη είναι το νέο καταστατικό που ρυθμίζει τα των ε, συνεργατών και βουλευτών. Οπότε, σήμερα χρησιμοποιούμε όλο όσο δικαιούμαστε. Άρα, αφού χρησιμοποιούμε όλο το χώρο μας, χρησιμοποιούμε και άλλο χώρο. Χρειάζονται επίση κάποιε εργασίε ώστε να φρεσκαριστούν κάποια κτίρια. Το, το, το παλιό παλιό το PHS και το Αλτιέρο Σπινέλη, το δεύτερο στη σειρά. Και επίση χρειαζόμαστε επομένω κάποιο μεταβατικό το σπιν ώστε όταν γίνονται οι επισκευέ να πάει εκεί ο κόσμο τον οποίο τα γραφεία επισκευάζονται. Και επομένω κρίνουμε ότι τώρα έχουμε αυτή την ευκαιρία για να αγοράσουμε ένα κτίριο κοντά στο Κοινοβούλιο και το ΤΡΕΒ έρχεται στην συνέχεια των, των κτηρίων ε, D4045. Επομένως, ε, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Βέβαια, η κατανομή αυτού του χώρου πρόκειται να προγραμματιστεί με κριτήρια αποτελεσματικότητας και ανάλογα και με την χρήση ε, στην οποία θα παραδοθεί το κτίριο. Οπότε θα πρέπει έτσι να δούμε ποια είναι η πιο δοκιμή λύση για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι δε λόγια του οποίου προτιμούμε την αγορά από την εκμίσθωση του γνωρίζετε. εξοικονόμηση χρημάτων μακροπρόθεσμα και επίσης πλεονεκτήματα ε, φορολογικά. Οπότε έτσι έχουμε καλύτερη διαχείριση του κτηρίου από πολλές πλευρές. Έχουμε επομένως την, ε, με αυτό το ότι τη σύμβαση των 99 ετών ε, μίσθωσης, συγχρονομίσθωση που θα καταλήξει σε οψιόν αγοράς Πρόκειται για ε, δημόσια σύμβαση που θα γίνει με αυτό το, το κτίριο στην Τρέβη και όπως προείπα και αυτή η λύση μας προσδίδει κάποια φορολογικά πλέον εκτίματα. Δεν έχουμε ε, ε, αμύαντο εκεί στο κτίριο αυτό, στη, στη Στρέβη, όπως ακριβώς ε, αποφασίστηκε και τον Ιανουάριο να εξεταστεί. Επομένως δεν έχουμε κανένα είδου κίνδυνο για την ε, ανθρώπινη υγεία με δεδομένη κάποια φυσιολογική χρήση, κάποιες εργασίες συντήρησης, επισκευές, ε, ούτε έρχεται σε αντίθεση με την υγειονομική νομοθεσία. Βεβαίω, όπως είπε ο κύριος Μπόρος, πέραν όλων αυτών θα ασκούμε τακτικούς ελέγχους όσον αφορά την ύπαρξη και συγκέντρωση ε, αμοιάντου. Επομένως, είμαστε σύντονοι με το ισχύον δίκαιο καθόλου. Η ιδέα αγορά των ακινήτων εδώ, στη, στη γειτονιά των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων, όχι μόνο δεν έχει πέσει κατά την ε, οικονομική κρίση, αλλά έχει γνωρίσει και κάποια άνοδο για λόγους προφανείς, διότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ζήτηση σε αυτή την ε, περιοχή των Βρυξελών για προφανείς λόγους και γι' αυτό και η εξέλιξη στην αγορά επίσης μας, ε, μας, μας, μας λέει ότι πρέπει τώρα να αγοράσουμε διότι στο μέλλον κατά τις προβλέψεις. Οι τιμές των ακινήτων εδώ, στο Cartier Leopold, το ευρωπαϊκό, Όλες οι τιμές λοιπόν δεν θα έχουν πέσει, αντιθέτως θα έχουν ανέβει. Και όπως ακούσαμε τον κύριο Λεβαντόσκη και τον κύριο Μπόκρος, ακούσαμε το ότι συμφωνούμε, συμφωνεί και το Προεδρείο, ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. σύμφωνα με τους ειδικού η τιμή κυμαίνεται στα λογικά επίπεδα που μπορεί κανείς να βρει ένα κινητό στην αγορά. «7.000 τετραγωνικά είναι το κτίριο. Καλό αυτό. Η θέση του κτίριου, η κατάσταση, η καλή του κτιρίου. Δεν θα χρειαστούν και πάρα πολλές ε, εργασίες. Και 2 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να εκταμιεύσουμε για τις εργασίες αυτές και όπως μας υπενθύμησε ο κύριος Μπόκρος έχουμε 22,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μεταφερθούν στην επόμενη χρήση για να τα δώσουμε στο βελγικό κράτος και τα υπόλοιπα θα βγουν από το αποθεματικό. Το Προεδρείο εξέθεσε όλες τις πληροφορίες σας στην Επιτροπή σας τον Οκτώβριο. Και επίσης την προηγούμενη εβδομάδα σας στείλαμε ακόμα περισσότερα στοιχεία. Οπότε το, το Προεδρείο θεωρεί ότι πρόκειται μια μοναδική ευκαιρία. Να μην τη χάσουμε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεπέδη. Κύριε Ολμάγερ, έχει το λόγο και μετά ο κύριος Σιγητής. Πρόεδρε, και εγώ νομίζω ότι είναι σωστό να αγοράσουμε μάλλον να ζητήσει από τον συνάδελφο από τους Δημοκράτε. Καλύτερα να αγοράσουμε και να μην νοικιάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Είμαι επιπισμένη ότι υπάρχει συμπληρωματική ανάγκη χώρου είναι σωστό. Μου φαίνεται επίση ότι είναι καλό που το κτίριο αυτό βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί μάλιστα να συνδεθεί άμεσα. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, θετικό. Αυτό που δεν μπορούμε να κρίνουμε είναι η κατάσταση ότι έχουμε μια τιμή 33% πάνω από τη τιμή αγορά. Δεν είναι πολύ εύκολο να το κατανοήσουμε. Αλλά αν δεν μπορεί κανένα εύκολα να επιλέξει βέβαια το κτίριο που θέλω, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Το ίδιο έχει γίνει νομίζω και με το κτίριο Eastman αυτό που, που λείπει όμως είναι η γενική εικόνα των κτίριων και των χώρων στο κτίριο. Δεν υπάρχει ακριβές οργανόγραμμα, δεν υπάρχει ε, ένας προγραμματισμός σφαιρικός που το έχει ζητήσει Πλιστάκη στο Κοινοβούλιο και μου φαίνεται αναγκαίο μακρο, βραχυπρόθεσμα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης για να μπορούμε να υιοθετήσουμε μακροπρόθεσμα ε, σχέδια. Και είμαι πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε περισσότερο λεπτομέρειες. Όσον αφορά τον αμύαντο όμως ανησυχώ. Όχι μόνο για την υγεία του προσωπικού, γιατί θα υπάρχουν συμπληρωματικά ε, ε, στην ανακαίνιση, γιατί η ανακαίνιση αυτή τη στιγμή θα κοστίσει περίπου 2,5 εκατομμύρια λέμε, αλλά ε, είδα σε πολλά κτίρια την κατάσταση με τον αμίαντο στη χώρα μου, ότι μετά από πέντε χρόνια περίπου υπάρχει τεράστια ανάγκη για πανάκριβο ε, πανάκριβη ανακαίνιση λόγω της ε, ε ύπαρξης και θα πρέπει να το πούμε αυτό στον πολιτή. Δεν μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος. Δεν ε, μπορεί κανένας να αγοράσει το βάρος του παρελθόνος και να πληρώσει και το 33% πάνω από την τιμή αγοράς. Θα πρέπει να υπάρχει μια ε, νομική εξασφάλιση, γιατί ακόμα και αν οι γνωμοδοτήσεις αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν είναι τόσο ψηλέ ε, οι πιέσει αυτές, είδα πολλά κτίρια που μετά από 5-10 χρόνια παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα ότι ο αμύαντος βγαίνει από το τσιμέντο, από το μπετόν. Και ένα τμήμα βγαίνει από τους, από τους αγωγούς ε, κλιματισμού. Και όπως λέγεται καμιά φορά θα πρέπει να κρεμίσει όλο το κτίριο. Ε, εντάξει, δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά πως θα είναι πανάκριβη η εξυγίανση και ανακαίνιση και όλα αυτά ε, στην πλάτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την τελευταία αναλύση του φορολογούμενου δεν μου φαίνεται ότι είναι καλό. Προβληματικό μου φαίνεται και θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να φροντίσουμε να υπάρχει μια νομική ασφάλεια. Δηλαδή καταρχήν είμαι υπέρ της αγοράς ε, του κτηρίου αλλά λυπούμε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν τηρήθηκε η συνεπής και ανοιχτή στάση έναντι του Κοινοβουλίου που το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε κατά βάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ιντιμπορκ. Ναι, για το θέμα αυτό του Αμιάντου. Θα ήθελα να αναφερθώ και εν ώψη της ιστορίας του Αμιάντου στο Στρασβούργο. Εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά νομικά θέματα αντιβρασμένη θητεία. Ανησυχώ λοιπόν ότι με το ίδιο πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα του Μιάντου στο Στρασβούργο, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το σημείο. Και αυτό το φλαματικό έγγραφο θα πρέπει να το διαβάσουμε. Προσεκτικά, εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά φλαματικά και ο αντιπρόεδρος φαντάζομαι όχι. Πώς ε, συμπληρωματικές διαπραγματεύσεις μπορούμε να κάνουμε. Τι γίνεται όσον αφορά την ευθύνη για το αμίαντο και είναι η εξασφάλιση από την ευθύνη αυτή καλύτερα από τη στο Γιατί α, το νομικό θέμα εξακολουθεί να είναι ανοιχτό στο Στρασβούργο. Θα θελήσω να με καθεσκάσετε, αλλά θα πρέπει να είναι σωστή η καθησύχαση αυτή. Στο παρελθόν ο συνάδελφος ε, Νέστα μιλούσε για άκακο αμίαντο. Μετά από ό,τι είχαμε τα προβλήματα, ξαφνικά ο αμίαντος ξανά πολύ επικίνδυνος. Δεν θέλω να ξαναζήσω τα ίδια. Πρώτα σας ευχαριστώ ο κύριος Γκάιερ και μετά θα σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ο κύριος Γκάιερ. Μια απλή ερώτηση προς τον κύριο Αντιπρόεδρο. Σε ποια μελέτη της αγοράς βασίζεται όταν λέει ότι αυξάνονται οι τιμές ε, των ε, ακινήτων στο, στην περιοχή αυτή της, ε, των ευρωπαϊκών κτηρίων. Εγώ έχω ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Λεπρόδος. Κατόπιν της συζήτηση αυτής, κύριε Σιγητά, τι μας προτείνετε. Thank you. the state of play is as follows. Σας ευχαριστώ. Η κατάσταση έχει ως εξής. Είναι μια απόφαση του Προεδρείου που ελήφθη τον Ιούνιο. Θετική σε σχέση με τα πρότυπα που ακολουθούμε. Η πρόβλεψη για τις τιμές των ακινήτων στις Βρυξέλλες τότε ήταν κάπως διαφορετική από τη σήμερα αλλά η σύγχρονη χρηματοπιστωτική λογιστική και η συναλλαγή αποφασίστηκε στο Προεδρείο. Εμείς θα πρέπει να αξιολογήσουμε την δημοσιονομική πτυχή της απόφασης, δεδομένων κάποιων επιφυλάξεων που εξακολουθούν υπάρχουν στην αίθουσα. Όλοι καταρχήν είναι υπέρ της αγοράς ενός νέου χώρου για το Κοινοβούλιο στην καλύτερη δυνατή τιμή αλλά οι επιφυλάξεις αφορούν και αυτό είναι και το μάθημα που αποκομίσαμε από το Στρασβουρού για τον αμύαντο και για τα προβλήματα και ίσως μια πιο ανεπτυγμένη σύγκριση προτύπων ε, δημοσιονομικής, ε, λογιστικής και η σε σχέση με τις διαφορετικές απόψεις και όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών ε, στην αγορά των Βρυξελών. Θα πρέπει να λάβουμε μια τελική απόφαση στην επόμενη συνεδρίασή μας που είναι νομίζω την 1η Δεκεμβρίου. Και εδώ μεταξύ εγώ μπορώ να σας προετοιμάσω σε περισσότερες επεξήγησεις, αλλά βασικά βλέπω να είμαστε υπέρ μετά από κάποιες ε, ακόμα επεξηγήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούκρος και μετά η κυρία Ντουιρά και μετά κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Εγώ δήλωσα ξεκάθαρα ότι καταρχήν είμαι υπέρ της αγοράς αυτής. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει καμιά παρεξήγηση περί αυτού. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω προ όφελο ολόκληρη Επιτροπής ότι δεν είναι καλό να έχουμε περιστασιακή ενημέρωση που θα μας στάνει μόνο μετά από πολλή πίεση. Ο κύριος Αντιπρόεδρος είπε και σήμερα πως το κτίριο δεν έχει αμίαντο. Μα δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Όχι, δεν είναι ούτε καν ασφαλές. Αν διαβάσετε το φλαμαδικό κείμενο, το έκαναμε. Διαβάσαμε το κείμενο. Το ζητήσαμε αυτό και την περασμένη φορά, αλλά πολύ αργά μας έφτασε. Όταν έφτασε το έγγραφο αυτό ήταν ατελές. Οι σελίδες που έλειπαν έφτασαν μόλις σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί. Και εκεί ανακαλύψαμε πώς πραγματικά είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Υπάρχουν ωστόσο διάφοροι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε και πάλι τονίζω, εγώ δεν θέλω να τορπιλήσω αυτή την αγορά, αλλά είναι υποχρέωση αυτής της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι η, ε, το, το θέμα της ασφάλειας του κτηρίου θα μπει στο νομικό κείμενο και ως συνέπεια μπορεί ή να μην ε, ή μπορεί και όχι να έχει επίπτωση στην ε, τιμή αγοράς ή στον κόστος ανανοικοδόμησης ή, ανα... ή ε, διόρθωσης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε μόνο τις οικονομικές επιπτώσεις χωρίς να λάβουμε υπόψη τίποτα άλλο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσέξουμε όλες τις πτυχές ταυτόχρονα. Μπορούμε να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα θέματα σύντομα. Σε αυτό συμφωνώ με τον Γιάννου Λεβαντόφσκι ότι πιθανότητα όλη αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει μέσα στο μήνα και να ψηφίσουμε την 1η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λιωγό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. Άκουσα όλες τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις που έλεγχαν. Είναι νομίζω νόμιμο, είναι λογικό να αναρωτιέται κανένας για το χώρο που προσφέρεται το αναμίαντο κλπ. Είναι νομίζω πολύ νόμο που αναρωτιέται τα πράγματα αυτά η Κομισιόν. Πήραμε νομίζω πολλέ από τι απαντήσει και ιδίω όσον αφορά τον χώρο, το συζητήσαμε και στο Προεδρείο αυτό. Και απολύτω την κυρία εκεί που ρώτησε, είναι δύσκολο να πούμε ότι υπάρχουν τόσε θέσει ε, απασχόληση και τόσα τετραγωνικά και έτσι καλύπτονται οι ανάγκε. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλέ θέσει. Ε, που, ανθρώπων που έρχονται ε, για μια μέρα την εβδομάδα, άλλο που είναι πέντε μέρε την εβδομάδα, άλλο που είναι μαθητεμόμενοι άλλο που έρχονται για λίγο χρονικό διάστημα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ ευέλικτοι και να εξάσουμε τα πράγματα με προσωμείωση και δεν μπορούμε να είμαστε ακριβεί σε ένα τετραγωνικό. Όσον αφορά το θέμα τη ε, μελέτη αγορά και των μελετών που λένε ότι υπάρχουν πολλά άδεια γραφεία στις Βρυξέλλες, ε, αλλά μπορώ να σα εγγυηθώ ότι στο Ευρωπαϊκό ε, στην ευρωπαϊκή εδώ γειτονιά η τιμή αυξάνεται με προοπτική αύξησης ανά τετραγωνικό ή ένα γραφείο. Και γι' αυτό η πρόθεση να αγοράσουμε είναι μια πρόθεση για να περιορίσουμε για το Κοινοβούλιο μακροπρόθεσμα τις δαπάνε. Και τρίτο για το αμίαντο, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καθησυχαστούμε, γιατί καταλαβαίνω ότι το, ε, σοκ ήταν πολύ μεγάλο για το Στρασβούργο. Είναι νομίζω νόμιμο τον ρωτάτε και θα έχουμε ε, απαντήσεις ε, έγκαιρα. Πραγματικά ήταν κάπως καθυστερισμένο να πάρετε την έκθεση αυτή για το... στο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ όμως που το διαβάσατε και επιστήρετε την προσοχή μας σε κάποια σημεία που επιτρέπουν αυτό όλο να γίνει με τις καλύτερες εγγύσεις κατά από τους καλύτερους όρους. όλων φυσικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία Λιγό που ξέρουμε ότι, μπορεί, ότι διαβάζει φλαμαδικά. Ο κ. πρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όσον αφορά την τιμή, το τίμημα, το λέμε Βαλέρ Βένα. και είναι 22,6 εκατομμύρια. Όμως, θα πρέπει να προσθέσουμε ένα 32% και κάτι διότι δεν θα γίνει πώληση με δημοπρασία. Άρα άλλο είναι η βασική τιμή και άλλο είναι αυτό. Διότι θα έχουμε αυτή την προσάυξη του 33%. Άρα 31, κάτι της εκατό είναι η τιμή της αγοράς. Και εν πάση περιπτώσει, κινούμεθα στα πλαίσια των, των τιμών των αγορέων, δεν είναι φουσκωμένη τιμή. Ε, διότι εδώ, σε αυτή την περιοχή των Βρυξελών που είναι τα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με αυτά που μας λένε επαγγελματίε του κλάδου, μεσίτες, Κατά το δεύτερο τρίμηνο η αγορά αναθερμάνθηκε έφτασαν να έχουμε και αυξήσεις μέχρι και 6% σε μερικές περιπτώσεις. Άρα δεν έχουμε καμία πτώση των τιμών, ειδικά σε αυτή την περιοχή των Βρυξελών, διότι η ζήτηση παραμένει έντονη. Τώρα, όσον αφορά τον αμύαντο, σύμφωνα με την ενισχύει νομοθεσία, το κτίριο χαρακτηρίζεται ως ασφαλές από πλευράς αμύντος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να υπάρχει αμύντος που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. Και ο αμύδος που είναι κάπου παγιδευμένος στο χώρο σημαίνει ότι η περιεκτικότητα στην ατμόσφαιρα του κτίριου είναι στα πλαίσια τα επιτρεπόμενα από την ε, υγειονομική νομοθεσία. Έτσι έχει κατάσταση σήμερα. Πέραν αυτό τώρα, Πρόεδρε. Περιοριζόμαστε μια προθεσμία που είναι η 30 Νοεμβρίου. Εάν δεν απαντήσουμε με τρόπο αοριστικό ή στον πολιτή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα χάσουμε την ευκαιρία. Οπότε, εάν έχουμε αναβολή, τότε υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος ε, να χαθεί η ευκαιρία ή θα χαθεί και σίγουρα. Ε, euh, Ωραία, σας ευχαριστώ. Ο κ. Σιγηρής έκανε μια πρόταση. Ναι, ναι, το ίδιο όπως πριν. Υπό όρους, ναι. Και αυτό μπορεί να μεταβληθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η, πρώτη δόση να πληρωθεί τέλη Νοεμβρίου. Και νομίζω ότι αν υπάρχει μια μέρα καθυστέρηση δεν θα είναι και τραγικό. Αυτή την εντύπωση έχω. Υπό όρους. έχουμε πολλές επιφυλάξεις. Κανένας δεν ε, αμφιβάλλει για τις, ε, τις πηγές των πληροφοριών που έχουμε. Αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις. Θετικά διακείμενοι όσον αφορά την αγορά, αλλά επιφυλάξεις όσον αφορά αυτές τις παρατηρήσεις που έγιναν, απαντήθηκε μέρος από τον αντιπρόεδρο, δηλαδή οι πόρους ναι προς τον πολιτή και ψηφοφορία στι 1η Δεκεμβρίου. Βέβαια, εσείς κύριε Πρόεδρε μπορείτε να θέλετε να ψηφίσετε τώρα αμέσω. Αυτή η σύστασή εσει κυριε είναι πάντως. Πρόεδρος, ευχαριστώ Σεμφαντόρ. Εάν η συσταση μου ειναι παντω ευχαριστω είναι 30 Νοεμβρίου, τι θα γίνει. Την οποία εμεί είμαστε εκπρόθεσμοι σε Παρίσι, Μαδρίτη, κάπου αλλού. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει αν εμεί ψηφίσουμε την πρώτη του μηνό. Ε, αφού θα έχει εκπνεύσει η προθεσμία το τότε, τότε θα ισχύει διαφορετικό νομικό και θα πρέπει αυτό να έχει ξεκαθαριστεί. Και εγώ ψηφίζω επομένω σήμερα να ψηφίζω για να μην περιμένω μέχρι, μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών και έτσι έχουμε αυτό το οποίο μας είπε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, ο κ. Αντιπρόεδρος, ναι, ε, νομίζω ότι η τιμή είναι σαφής και όσον αφορά σε σχέση με την ε, τιμή αγοράς ε, και όσον αφορά την εξέλιξη αγοράς, αυτό είναι σαφές. Το μόνο σημείο που παραμένει κάπως ανοιχτό είναι το θέμα του αμοιάντου. Και όπως σας είπα, μπορούμε να αγοράσουμε το κτίριο όντα σίγουροι ότι είναι σύμφωνο με τη σημερινή νομοθεσία για τον αμίαντο. Αυτέ είναι οι πληροφορίε που μπορώ να σα δώσω. Είναι ασφαλές όσον αφορά τον αμίαντο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας δώσετε το πράσινο γιατί 30 Νοεμβρίου είναι η καταλλακτική προθεσμία. Και άμα μου λέτε τώρα θέλει να ψηφίσετε την 1η Δεκεμβρίου, είναι σαν να λέτε ότι θα χάσουμε την ευκαιρία που θα είχαμε. Ο εισηγητή. Να τροποποιήσω την πρότασή μου. Υπό το βάρος των ε, επιχειρημάτων του συντονιστή και του κυρίου Αντιπρόεδρου μπορούμε σήμερα να αποφασίσουμε υπό τον όρο ότι πριν από 30 Νοεμβρίου θα λάβουμε γραπτές εξηγήσει όσον αφορά το θέμα αυτό του αμοιάντου και το θέμα της ευθύνης. Αντίστροφα δηλαδή. Πρόεδρος, ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Γιατί τώρα μια μισή ώρα εξετάζουμε το θέμα αυτό για 30 εκατομμύρια. Και έχουμε μια μισή ώρα διαπραγματευτεί για 136 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, προτείνω να ψηφίσουμε πάνω στην πρόταση του δηλαδή να δώσουμε το πράσινο φως για την πληρωμή υπό τον όρο ότι πριν από τις 30 Νοεμβρίου 30, 30, 30 Νοεμβρίου, ναι το Προεδρείο θα μας δώσει όλες τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τους εισηγητής και όσον αφορά για τον τρόπο υπολογισμού της τιμής και όσον αφορά τον αμίαντο. Ποιο είναι υπέσπρο της αυτής. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Attention de M. Bocros au groupe et du groupe socialiste et du μια ε, πλειοψηφία υπέρ αποφασίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, περνάει η ώρα. Εμείς δεν μπορούμε να σταματάμε τώρα λόγω σε όλα τα θέματα. Επανερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 6. Θα πάμε πολύ γλίγορα. Σημείο 6. Είναι γνωμοδότηση γνωμοδότηση Επιτροπής Προπολογισμών προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για την πρόταση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση χρηματοδοτικού μέσου για συνεργασία με τι εκβιομηχανισμένε χώρε. Είχαμε τη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Είμαι εισηγητή. Και έχουμε. Λάβει μία τροπολογία επαρίθμων 4 που προσθέσει στην τροπολογία 3. Μια τροπολογία που έχω εγώ, εγώ προετοιμάσει. Α, ωραία. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Εγώ είμαι ο εισηγητής. Κατά. Ποιος τολμάει να είναι αντίθετος. Αποχές, δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται, ευχαριστώ. Τροπολογία 2 που έχω υποβάλει. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία. Αποχές. Ένα κατά μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 3. ίδια πλειοψηφία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Του κ. Καλτιέρη. Εγώ δεν είμαι υπέρ γιατί δεν είναι σύμφωνη η τροπολογία με την αρχή που ακολουθούμε συνήθως εδώ. Ποιος είναι υπέρ. Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Α, για, για, για να μετρήσουμε. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, ça suffit. Euh, pardon, 15. <laughs> Qui est con 15. Κατά. Ποιος είναι κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et il y a une, une abstention, si je comprends. Και μία εποχή από κατάλαβα. Οι φιλελεύθεροι Λοιπόν, 17 κατά δεν εγκρίνεται λοιπόν. Από εκεί και πέρα, για την πρόταση γνωματότηση ποιος είναι υπέρ, κατά, Κανένας αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 7. Ευρωπαϊκό Όρος Εθελοντισμού. Έχουμε μια γνωμοδότηση της Περμπαραματέρα και την οποία επίσης τελευταία φορά κάναμε τη συζήτηση. Μπορούμε αμέσως να περάσουμε λοιπόν στην εξαρτησία των τροπολογιών. Τροπολογία 7 της κυρία Βαλσάνη. Η συγκέντρια. Δεν ε, βλέπω τι προτείνει ο εισηγητής. Η συγκέντρια είναι κατά μου λένε, έτσι. Πριν Στη ψηφοφορία, Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι. Όσον αφορά αυτό το σχέδιο χνομοδότηση, εγώ ήθελα να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικέ πτυχέ. Η πρώτη αφορά την αύξηση του κονδυλίου, το νούμερο δηλαδή που δίνει η Κομισιόν και δεύτερον ποσοστό συγχρηματοδότηση. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, η Επιτροπή προέβλεψε 3 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις δράσεις προετοιμασίας για το 2011 και 6 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις ίδιες τις δράσεις του έτους εθελοντισμού που θα είναι το 2011. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, προπολογισμού εγώ πρότεινα μια αύξηση του κονδυλίου που πρότεινε η Κομισιόν. Και μάλιστα υπήρξε συνένεση από πλευρά άλλων συναδέλφων από άλλε πολιτικέ ομάδες όπως ε, οι σοσιαλιστές και άρα λοιπόν ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία που είχε σχέση με την αύξηση από 6 σε 8 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το κονδύλι. Και όσον αφορά ε, το τη δεύτερη παρατήρηση, εγώ αποσύρω τις δύο τροπολογίες, 5 και 6, που αφορούν ε, την ε, μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο, από το 80% στο 65% και γι' αυτό συμφωνεί και ο εισηγητής της Επιτροπής Πολιτισμού. Okay. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία εισηγητρία. Λοιπόν, οι τροπολογίες 5 και 6 έχουν αποσυρθεί και αν κατάλαβα σωστά η τροπολογία 10 έχει υποστεί μια προφορική τροπολογία για να περάσει σε 8 εκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα τις τροπολογίες που απομένουν με τη σειρά Άρθρο 2 παράγραφος 3 τροπολογία υπαριθμών 8 της κυρίας Μπαλζάνη. Η συγχύτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Για να μετρήσουμε. Les gros bataillons de la gauche sont Je remercie. 13 υπέρ. Κατά. <laughs> Je pense que Les contre sont plus nombreux. Μάλλον κατά είναι πιο πολύ. Αποχές. Καμία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 9 της κυρίας Μπαζάνη. Η ίδια κατάσταση η εισηγείται είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Οι ίδιες πλειοψηφίες. Ευχαριστώ. Κατά. Ναι, το ίδιο. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 10 με την προφορική τροπολογία της κυρίας Ματέρα. Υπέρ, κατά, μία ψήφος κατά. Αποχές, εγκρίνεται λοιπόν, με μία αποχή. Όπως το επιπήθηκε από την κυρία Ματέρα. Τροπολογία 3 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας. που είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 5 και 6 έχουν απορριφθεί, ε, αποσυρθεί και έχουμε μετά τροπολογίες κυρίας Παρζάνη. Να τις πάρουμε όλες μαζί τις τροπολογίες αυτές. Α, ναι. 11, 12, 13 και 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία κατά της κυρίας Βαρζάνη που είχαμε και προηγουμένως. Αποχές. Απορρίδονται λοιπόν. Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Παράγραφό στον 1α, νέο. Τροπολογία 1 της εισήγητες. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Η αριστερά είναι κατά. αποχε Η απλή λοιπόν. Και για το 2 φαντάζομαι το ίδιο γίνεται. Όχι, τροπολογία 2, μεγάλη πλειοψηφία. Κατά, αποχέ. οι δύο τροπολογίες αυτές συγκρίνονται. Τέλος. Για το τροποποιημένο μεθοδικό ψήφισμα υπέρ. Κατά. Ποιος τολμάει. Ένας κατά. Άποχες. Άρα. Κυρία Ματέρα, ομόφωνα, μείον ένα. Σας συγχαίρομαι. Χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή Πολιτισμού της Ουσίας Αρμόδια θα ψηφίσει 23 Νοεμβρίου και στην Ομέλεια 14 με 17 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ κύριε Συγγετρία. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8. Κύριε Χάουκ. Πήγαμε στη Ιούτα. Ja, da gibt's ja etliche. Nee. Ναι. Υπάρχουν πολλές μεταφορές εδώ. Εν μέρη παλιές, εν μέρη καινούργιες. Για να αρχίσουμε με εκείνες που ήταν πολύ ήπιο μέχρι περασμένη εβδομάδα. Είναι η 35 για τη Ζανχάη. και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Έκθεση Σανγκάη. μερασμένη συνεδρία της Επιτροπής μας είχαν υποβάλει μια σειρά ερωτήσεων. Πήραμε πέντε σελίδες γραπτή απάντηση από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Εγώ ικανοποιήθηκα από τις απαντήσεις αυτές, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά η Κομισιόν πραγματικά απάντησε πάρα πολύ αναλυτικά με σκίτσα και με όλα ότι χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε περί τίνους πρόκειται και τι πρόκειται η Κομισιόν να κάνει με τα χρήματα αυτά τα οποία θα τις χορηγηθούν. Εάν δεν υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις και όλοι οι συνάδελφοι έχουν ικανοποιηθεί και θεωρούν ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες για το έτσι αυτή μεταφοράς, προτείνω στους συναδέλφους να ψηφίσουμε υπέρ. Πράγματι, πολύ ωραία. Πραγματικά συζητήσαμε αναλυτικά το θέμα την προηγούμενη φορά. Ποιο είναι λοιπόν υπέρ τη μεταφορά αυτή που προτείνει η συγγετρία. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχέ. Μεταφορά 35. Εγκρίνεται λοιπόν. 40. Ναι, στο 40 λέμε ότι θα πρέπει να άρουμε το αποθεματικό για την ΕΦΣΑ στην Πάρμα. Το είχαμε να βάλει την περασμένη φορά γιατί δεν είχαμε ακόμα την απάντηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά πόσο η Επιτροπή αυτή είναι υπέρ ή όχι. Εν τω μεταξύ έχουμε μια θετική απάντηση. Προτείνω λοιπόν στους συναδέλφους να εγκρίνουμε τη μεταφορά αυτή. Πρόεδρος ευχαριστώ. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν. Και η μεταφορά 40. 43 τώρα. Αυτό πρόκειται για σχέδια ενέργειας. Ε, δίκτυα συλλογή ε, άθρακα και ε, σχέδια offshore γιατί από το διοικητικό τμήμα έχουμε κάποια χρήματα που περισσεύουν που δεν τα χρειάζεται η Κομισιόν και γι' αυτό μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε αυτά τα σχέδια. Την περασμένη φορά είχα ρωτήσει και ίσως μπορεί πολύ γλυγόρα να απαντήσει τώρα η Κομισιόν. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια, υπάρχει ένας κατάλογος με τα σχέδια αυτά, έχουν εγκριθεί. Μπορείτε να μας το δώσετε και αργότερα γραπτά. Απλώς απορώ. Με ενδιαφέρει. Γιατί όλους μας ενδιαφέρει νομίζω. Γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει γλίγορα τα χρήματα να δαπανηθούν από το σχέδιο ανάκαμψη. αν πρόκειται να υπάρχει θετικός αντίκτυπος στην εξυγίανση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να συμφωνήσουμε με τη μεταφορά αυτή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε για το 2009. Έτσι, ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Η μεταφορά 44. πρόκειται να αυξηθούν τα ε, το πρόγραμμα για τις μελέτες. Οι μελέτες αυτές, λέει η Κομισιόν, χρειάζονται για να μπορέσει το πρόγραμμα στο χωρο 2010 2010-2014 να πραγματοποιηθεί σωστά. για να μπορέσει το νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν να προχωρήσει όπως πρέπει. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δώσουμε στις Κομισιόν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής. Κατά. Μία ψήφος κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 45. Πάλι πρόκειται για διοικητικό δαπάνε για προσωπικό που δεν χρειαστήκε γιατί δεν μπορούσε να γίνει το χρυσόγραφα προσλήψης. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα που πέρισεψαν και μπορούν να δοθούν για το σχέδιο Γαλιλαίο. Και μπορούμε παρά να είμαστε υπέρ, παρά να, εξαφανιστούν τα κονδύλια αυτά κάπου, καλύτερα να τα πεθούν σωστά. Πρώτα, σταυμάσια. Ζήτω ο Γαλιλαίος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μεταφορά 48 θα ήθελα να αναβάλουμε, Πρόεδρε, μέχρι να συζητήσουμε την έκθεση του Ράιμερ στο σημείο 11. Γιατί πάλι πρόκειται να δαπανηθούν κάποια χρήματα για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, θα έλεγα να αναβάλουμε, να περάσουμε στο 51 τώρα πρώτα. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν την έκθεση του Ράιμερ, τη δυναμική βάση. 51 η Πρόκειται για τη μεταφορά για τη Γεωργία, Γάζα και Κωσυφοπαίδιο. Μια αποστολή παρατηρητών στην Γεωργία όπου χρειάζονται πολλά τεθωρακισμένα οχήματα κλπ. κλπ. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε πολλές ερωτήσεις ίσως, αλλά νομίζω ότι αν θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους που ε, εκπροσωπούν την Επιτροπή Πολιτισμού στην αρμόδια επιτροπή. Δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα σε πνευματικέ ερωτήσει. Εγώ είμαι υπέρ τη μεταφορά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Συνήθω είναι πιο φτηνή η ειρήνη από ότι το πόλεμο. Ποιο θέλει να χρηματοδοτήσουμε την ειρήνη. Ποιοι είναι υπέρ τη μεταφορά αυτή, παρακαλώ, 51. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ πολύ. 52. Συγγνώμη. Α, από εκεί, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Απέχεται πάνω στην ειρήνη, ε. Λοιπόν, η ευφύης ενέργεια. Να δούμε, η πράσινη είναι υπέρ της ευφυούς ενέργειας. Ναι, θαυμάσια είναι όλα αυτά. Δυστυχώς δεν βρήκαμε αρκετούς που θέλανε να διαχειριστούν αυτή την ευφύ ενέργεια. Και γι' αυτό στην εκτελεστική υπηρεσία υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα που λέγεται τώρα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα ίδια τα σχέδια έλαβε χώρα ένα διαγωνισμό και υπευλήθηκαν πάρα πολλέ αιτήσει για προγράμματα, για σχέδια συγκεκριμένα και γι' αυτό θα μπορούσαμε αυτά τα 515.000 ευρώ να χρησιμοποιηθούν για άλλα σχέδια και όχι για προσωπικό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω. Πρόεδρος, ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής 52. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελευταίο μεταφορά. Όχι, πρώτη τελευταία μεταφορά. 54. Για τα ΜΜΕ. Το ίδιο. Το ίδιο είναι και εδώ σε άλλο τομέα της πολιτικής. Η εκτελεστική υπηρεσία δεν χρειάστηκε όλα τα χρήματα που προβλέπονται και γι' αυτό μπορούμε τώρα τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για τα ίδια τα σχέδια και δεν μπορώ παρά να προτείνω να συμφωνήσουμε με αυτή την πρόταση. Πρώτα σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής, με, όπως προτείνει η συγκήτρια. Κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Ένας κατά εγκρίνεται. Τέλος. 55. Ιδέες λέγει. Το ίδιο πάλι η εκτελεστική υπηρεσία η οποία εργάζεται για να βοηθήσει το Συμβούλιο Έρευνας δεν προσέλαβε όσο προσωπικό είχε προβλέψει αρχικά. Ίσως δεν χρειαζόντουσαν τόσο προσωπικό και τα χρήματα που υπάρχουν τώρα εκεί θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για τα ίδια τα σχέδια. Θα ήταν πολύ ευφύες νομίζω, γιατί ακριβώς το Συμβούλιο αυτό έρευνας θα πρέπει να διαχειρίζεται αυτά τα σχέδια μέσα στα πλαίσια του εβδόμου προγράμματος πλαίσιο. Θα παραμείνουμε στον ίδιο τομέα. Είμαι υπέρ λοιπόν να κάνουμε τη μεταφορά αυτή. Θαυμάσια, θαυμάσια μεταφορά. Από διοικητικό κόστος χρηματοδοτούμε τις ιδέες. τι ωραίο. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής. Ευχαριστώ, κατά. Ευχαριστώ, αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Και ευχαριστώ και συγχαίρω την Γιούτα Χάουκ. Επανέρχεται ο Γιάννης Λεβαντόφσκι και τον ευχαριστώ που δέχτηκε να ξανασυζητήσουμε το δικό του θέμα. Είμαστε λοιπόν, ναι ναι, αυτό ήταν το 9 και όχι, το 21 το αποσύρθηκε και να μας το εξήγησε. Λοιπόν, Επιτροπή των Περιφερειών, ΕΝΦ 5. Μήπως να αρχίσουμε με το δικαστήριο. Αυτή είναι η σειρά. Ναι, δικαστήριο. Δηλαδή 6, 7, 8 και 9. Συλλογική κινητοποίηση πιστώσεων ώστε να γίνει μια προκαταβολική πληρωμή 5 εκατομμύριων ευρώ για το νέο σύνολο κτίριων. Leasing μέχρι το 2026 προς το κράτος του Λουξεμβούργου. 2007 και 2008 επιτρέψαμε αυτή την προκαταβολή ώστε να μειωθεί το μελλοντικό φόρτο. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς δεδομένου ότι το πλεόνασμα για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι πιστώσεις εξευρέθη μέσω τη αμοιβή προσωπικού. αυτό θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τα όσα έχουμε συμφωνήσει το 2007 και 2008, δηλαδή προκαταβολική πληρωμή, καταβολή, ώστε να μειωθεί το μελλοντικό, ο μελλοντικός φόρτος. Είστε υπέρ, κύριε Σιγητά. Πρόκειται για τέσσερις μεταφορές. Μάλιστα, ψηφίζουμε συνολικά. Ναι, είναι για να, γίνουν, για να δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τέσσερις διαφορετικές πηγές. Είναι μία μεταφορά για μένα, αλλά βεβαίω. εντάξει, είναι τέσσερι. Αν μπλοκ ψηφίζουμε. Ναι, η γραμμή που τα παίρνει είναι μία, αλλά οι δωρητέ είναι τέσσερι. Μία ψηφοφορία unblock. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν αυτή τη μεταφορά που συστήνει ο ε, εισηγητής μας για το δικαστήριο υπέρ κατά τρεις κατά αποχές. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο Επιτροπή των Περιφερειών. Ναι. Είναι το INF ε, 5. Ε, Εδώ έχω κάποιο πρόβλημα. Η πολιτική για την αντικατάσταση προσωπικών υπολογιστών πρόκειται για 300.000 ευρώ. Είναι μια πολιτική των θεσμικών οργάνων είναι το ίδιο για την Επιτροπή των Περιφερειών και για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να προσπαθούμε να αντικαθιστούμε το 1 τέταρτο των προσωπικών υπολογιστών ετησίω. Ωστόσο, αυτό δεν είχε προβλεφθεί για το 2009 και χρειάζεται αιτιολόγηση. Είναι τμήμα μια μεταφορά. Επιτροπή των Περιφερειών και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Χρειάζεται πολύ καλύτερη αιτιολόγηση για τη μεταφορά ε, κονδυλίων στην αντικατάσταση των προσωπικών υπολογιστών. Εγώ υποστηρίζω το υπόλοιπο κομμάτι της μεταφοράς για την Επιτροπή των Περιφερειών. Είμαι κατά της αποδοχής σήμερα, θέλω να περισσότερες αιτιολογήσεις, για τις 289.000 ευρώ για την αντικατάσταση προσωπικών υπολογιστών υπέρ του υπολείπου. Δηλαδή, νέα τεχνική πλατφόρμα, τα υπόλοιπα κομμάτια ναι, επί, έπιπλα λοιπά. Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά κύριε Σιγητά λοιπόν, κάντε την ίδια πρόταση για δύο σχέδια μεταφοράς που έχουν τον ίδιο αντικείμενο αλλά αφορούν δύο διαφορετικά όργανα με την ίδια πολιτική, Επιτροπή Περιφερειών και Κοινωνική και Κοινωνική Επιτροπή. Και εδώ από την νομική άποψη πρέπει να πούμε να έχουμε αντίρρηση. Εσείς έχετε αντίρρηση λοιπόν σε κάθε μια από τις περιπτώσεις για το πρώτο τμήμα που είναι η αντικατάσταση των υπολογιστών. αλλά δεν έχετε αντίρρηση για τα υπόλοιπα. Τμήμα 2, 3 και 4. Προτείνεται να λάβουμε την ίδια απόφαση και για τις δύο επιτροπές, περιφερειών και κοινωνική και οικονομική. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε χώρια, γιατί είναι δύο διαφορετικά ε, θεσμικά όργανα. Λοιπόν, για την Επιτροπή των Περιφερειών ψηφίζουμε την πρόταση του εισηγητή, δηλαδή Αντίρρηση μόνο για το τμήμα 1, αντικατάσταση υπολογιστών. Όχι, Εγώ έχω αντιρρήσεις για την αντικατάσταση των υπολογιστών. Τέσσερα, ένα, α. Για το B και το C δεν έχω αντίρρηση. Αντίρρηση έχω μόνο για την εγκατάσταση των υπολογιστών. και αυτό γιατί δεν έχουμε ε, αρκετές, ε, αρκετή αιτιολόγηση. Και για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και εδώ είναι ξεκάθαρο. Αντικατάσταση είναι το 1, κεντρική ασφάλεια να έχουμε αντίρρηση για το 2. Μάλιστα. Επιτροπή Περιφερειών. Ο εισηγητής έχει αντίρρηση για το 1 α και όχι για το υπόλοιπο. Μόνο για το συγκεκριμένο σημείο. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη πρόταση του εισηγητή. σα Σας ευχαριστώ κατά αποχές. Μία αποχή. Αντίρρηση λοιπόν για αυτό το σημείο. Περνάμε τώρα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Και εδώ το ίδιο κύριε Ισίτα. Ακριβώς. Ένα. Μεταφορά για την αντικατάσταση υπολογιστών. Έχουμε αντίρρηση και ανάγκη για περαιτέρω αιτιολόγηση. Και το δύο. Κεντρική ασφάλεια και σύστημα ε, διοχέτευση είναι ε, ε, το ίδιο. Είναι οκ. Εντάξει λοιπόν, 2, 1. Αντικατάσταση προσωπικών υπολογιστών. Έχουμε αντίρρηση. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη αντίρρηση που είναι σύμμορφη με την προηγούμενη. Κατά. Αποχές. Τα ίδια. Σας ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη του κυρίου Λεβαντόφσκι. Ναι. Όχι. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα ακόμα σημείωμα από το ελεγκτικό συνέδριο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. για μετατροπή θέσεων AST σε θέσεις AD. Είναι το άρθρο 17 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Είναι μια μετατροπή που ε, οδηγεί σε, αποτα... σε χρημάτων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να το σημειώσουμε. Μάλιστα. Ωραία, δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση, άμα όλοι συμφωνείτε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι. Έχουμε ένα τελευταίο, μια τελευταία ψηφοφορία, το 10, σημείο 10, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Κυρία Πούλμαν, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι πιο απλό σε σχέση με αυτά τα οποία σύντησαν προηγουμένως, διότι εδώ έχουμε την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις ε, Χημικές Ουσίες του Ελσίνκη. Έχει 450 υπαλλήλου αυτή τη στιγμή αυτή η υπηρεσία και στεγάζεται σε ένα κτίριο 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Ωρα Προηγουμένω ήταν κυριότητα μια ασφαλιστική εταιρεία. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η υπηρεσία είναι ότι η υπηρεσία αυτή επεξεργάζεται εμπιστευτικά στοιχεία. Η εμπιστευτικότητα πολλές φορές είναι πολύ υψηλό επίπεδο. πρέπει πολλές φορές να έρχονται κάποια φορτηγά να φορτώσουν υλικό. Είναι επομένως ε, ε, εκεί που βρίσκεται και κάποιο κατάστημα και οπότε μπορεί να υπάρχει έλεγχο τη ασφάλεια. Οπότε λέμε ότι μπορεί να γίνει και εκεί μια χρονομίστοση. Μιλούμε για χώρο που πρέπει επομένως να καλυφθεί με κάποια σύμβαση 2.900 ε, μέτρων. Ακριβώς υπάρχει επομένω ανάγκη ασφαλείας και θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το άλλο κομμάτι του κτιρίου. 17,42 ευρώ είναι το κόστος τιμής των τετραγωνικών μέτρων ε, μαζί με την ανακαίνιση του κτίριου που θα πρέπει να γίνει. Άρα νομίζω ότι η τιμή είναι λογική. Εγώ, χωρίς καμία επιφύλαξη, προτείνω να εγκρίνουμε αυτή την ε, πρόταση, την πρόταση μίσθωσης. Έχει γίνει ανταλλαγή ε, ε, απόψεων την τελευταία φορά ε, με τον διευθυντή αυτή τη υπηρεσία. Δεν τον κουβάλισαμε και σήμερα. Επομένω, ποιοι είναι υπέρ τώρα, υπέρ τη πρόταση τη ιδρυά μα να μην υπάρξει ένσταση. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Συνάδελφε. τελείωσε η συνεδρίαση. Α, έχουμε και ένα άλλο σημείο. Ο Χάιμερ έχει συντάξει μια έκθεση όσον αφορά την κινητοποίηση αυτού του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για διάφορα θέματα. Όμως ε, ακόμη δεν έχει χειρομοδοτήσει η Επιτροπή Απασχόλησης. Ίσως θα πρέπει αυτό να αναβληθεί, να μην το ζητούμε σήμερα. Ναι, Πρόεδρε. Όντως, Συζητήσαμε την πρόταση Κομισιόν για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Ε, είχαμε βοηθήσει, είπαμε, την ε, Ολλανδία, την, ε, τη Βόλβο, την Αυστρία, 15, για 15 εκατομμύρια. Στη τελευταία συνάντηση η Κομισιόν δέχθηκε ότι εν ώψη της ψηφοφορίας θα πρέπει να συζητηθούν τα επιμέρους θέματα χωριστά και όχι όλα μαζί. Θα θέλαμε εμείς μια αποστομένη διαδικασία, αλλά έτσι όπως έγινε, δεν θέλουμε όλα να τα βάλουμε μαζί, γιατί μπορεί από τις, ε, κάποιες από τις περιπτώσεις χρηματοδότησης να είναι πιο περίπλοκη από τις άλλες. Η Γιούτα θα συνεργαστεί μαζί μου και έχουμε την γνωμοδοσία της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά θα ήθελα και άλλες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν μας ικανοποιήσει τότε θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τις παραγράφους 1 έως 4 της ε, έκθεσης. Ε, το 1 και το 2 αφορούν ε, την Volvo. Εκεί έχουμε υποβάλει κάποια ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράγραφος 3, Αυστρία. η Επιτροπή Απασχόλησης είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι μέτρα στήριξης μπορεί να ληφθούν. 6.500 ευρώ ανεργαζόμενος στην Σουηδία και 14.300 ε, θέσεις εργασίας έχουν χαθεί. Άρα εδώ έχουμε μια διαφορά όσον αφορά την ε, αποζημίωση για πόλη θέσεων εργασίας. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πρέπει να μας τα δικαιολογήσει η Κομισιόν. Έχουμε και την Heymans, μια εταιρεία Ολλανδική. Μας πει και εδώ η Κομισιόν τι γίνεται. Γιατί την πρώτη εταιρεία που έχει και θηγατρικές σε Βέλγιο και Μεγάλη Βρετανία. Άρα θα πρέπει να μας πει συνολικά τη θέση σε εργασίες έχουν χαθεί. Για αυτά τα μέτρα δεν παρέχει επαρκές δικαιολογίες η Κομισιόν. Δεν είναι αρκετό αυτό που μα είπαν ότι είναι σαν τι δράσει συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γενικού Ταμείου. Αυτό μα είπε δεν μα αρκεί. Πρέπει να μα τα πει η Κομισιόν αυτά κάποια στιγμή. ούτω ώστε να μπορέσω στο κείμενό μου να περιλάβω και τα όσα έχει πει η Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά να δω και τα σχόλια της ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Επειδή δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα, αλλά βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τα ερωτήματά σας που συγκεντρώνουν τα βασικά ερωτήματα της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και άρα περιμένουμε ε, τις απαντήσεις της γραπτός πριν από τη δική σας ε, έκθεση και πριν από την ψηφοφορία. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, και με την Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε οι εκθέσει αυτέ να μα παρουσιάζονται μία προ μία για να μην χρειάζεται να καθαριστερούμε όπω πρόσφατα έγινε με την Ευρωπαϊκή υπόθεση για ευνοϊκέ αποφάσει μόνο και μόνο επειδή αυτό είχε καθυστερήσει λόγω της Ιρλανδικής, του Ιρλανδικού φακέλου επί του οποίου είχαμε επιφυλάξει. Να θυμίσω ότι η επόμενη μα συνεδρίαση είναι την 3η 1 Δεκεμβρίου και την 4η 2 Δεκεμβρίου και η συνδιαλλαγή για όσους θα έρθουν είναι την Τετάρτη 18. Πριν χωρίσουμε όμως να ευχαριστήσω την ε, βοηθό Πάιβι Όμαν που είναι εδώ παρούσα. Ίσως πρέπει να σηκώσετε το χέρι, Αϊβή, να σας ε, δουν όλοι. Να τη χειροκροτήσουμε, διότι η Πάιβι συμμετέχει για τελευταία φορά σε αυτή την Επιτροπή Προπολογισμού. Είναι 8 χρόνια μαζί μας. Δεν θα μας εγκαταλείψει τελείως, διότι έχει προσληφθεί χάρη στις μεταφορές που εγκρίναμε την προσλαμβάνει ο οργανισμός των χημικών προϊόντων του Ελσίνκη και τουλάχιστον θα είναι κοντά στην οικογένειά της χωρίς να εγκαταλείψει το Ευρωκοινοβούλιο και θα έχουμε την ευκαιρία να πιούμε μια σαμπάνια για να την ευχαριστήσουμε και να γιορτάσουμε τη συνέχεια της σταδιοδρομίας της πέρα συνεδρίαση, θα τα πούμε στην συνδιαλλαγή. Bon,